η ομάδα ECR ανακοίνωσε στο κοινο... στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι ο κύριος Μάρκους Πρέτζελ δεν είναι πια μέλος αυτής της ομάδας από 12 Απριλίου του τρέχοντος έτους και ότι θα είναι πλέον μία γεγραμμένος βουλευτής.